για το 2013 και θέλω πρώτα να παρακαλέσω εξ ονόματος του Συμβουλίου τον Προεδρεύοντα Υπουργό Δημήτρη Κούρκουλα να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Εκ μέρους της Προεδρίας θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και κυρίως την κυρία Όμεν Ρούιτεν για το έργο της. Το ψήφισμα υπογραμμίζει μια σειρά θεμάτων και ανησυχιών βαρύνουσας σημασίας και έρχεται σε μια ιδιαίτερη χρονική συγκυρία για τις σχέσεις ευρωπαϊκής ένωσης τουρκίας. το συμβούλιο επιβεβαιώνει τη σημασία που αποδίδει στις σχέσεις της εε με την τουρκία. η τουρκία αποτελεί για την εε τόσο μια υποψήφια χώρα όσο και ένα σημαντικό εταίρο με δυναμική οικονομία οι ενεργές και αξιόπιστες συνταξιακές διαπραγματεύσεις βασισμένες στην καθιερωμένη αιρεσιμότητα θα προσδώσουν στη σχέση αυτή με την τουρκία την πλήρη δυναμική τους. στο πλαίσιο αυτό χαιρετίζουμε το άνοιγμα πέρσι του κεφαλαίου 22 περιφερειακή πολιτική και συντονισμός διαφορετικών μέσων. η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να παραμείνει ο καταλύτης για τις μεταρρυθμίσεις στην τουρκία ειδικά στους τομείς του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών. το συμβούλιο συνεχίζει να ενθαρρύνει την τουρκία να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα παρέχουν τις απαραίτητες δικλείδες ελέγχων και ισορροπιών εξασφαλίζοντας ελευθερία δημοκρατία ισότητα κράτος δικαίου σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητε. η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων βάσει των ευρωπαϊκών κριτηρίων αποτελεί ζήτημα κομβικής σημασίας. το συμβούλιο επίσης σημειώνει θετικά την ενεργό και συνεχώς αναπτυσσόμενη κοινωνία των πολιτών στην τουρκία η οποία θα πρέπει να υποστηρίζεται και να ενθαρρύνεται ως παράγοντας που διαθέτει νομιμοποίηση. το συμβούλιο εξάλλου χαιρετίζει άλλες σημαντικές θετικές εξελίξεις μεταξύ των οποίων την δημιουργία και την έναρξη λειτουργίας θεσμών όπως ο συνήγορος του πολίτη η εθνική αρχή για τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί στον τομέα των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων. εντούτοις περισσότερες και συνεχείς προσπάθειες θα χρειαστούν ειδικά όσον αφορά στη βελτίωση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών στην τουρκία τόσο στην νομοθεσία όσο και στην πράξη συμπεριλαμβανομένων των τομέων της ελευθερίας της έκφρασης της ελευθερίας του συναθρίζεσθε, της θρησκευτικής ελευθερίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων η υπερβολική χρήση βίας εναντίον διαδηλωτών από τα όργανα επιβολής του νόμου πρέπει να αντιμετωπίζεται και να διερευνάται αποτελεσματικά. οι πρακτικές περιορισμών στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης συμπεριλαμβανομένου μεγάλου αριθμού δικαστικών διώξεων κατά συγγραφέων και δημοσιογράφων ακαδημαϊκών και υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι συχνές και δυσανάλογες απαγορεύσεις ιστοτόπων websites καθώς και η ευρεία εφαρμογή της νομοθεσίας για την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα αποτελούν ζητήματα που επίσης εγείρουν σοβαρές ανησυχίες. επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ότι τα ζητήματα που προβληματίζουν την ευρωπαϊκή ένωση επισημάθηκαν στον πρωθυπουργό της τουρκίας κ. ερντογκάν κατά τις συναντήσεις που είχε με τους προέδρους βαν ρομπόι μπαρόσο και σούλτς κατά την επίσκεψή τους στις 20 ιανουαρίου στις βρυξέλλες. οι πρόεδροι βαν ρομπόι και μπαρόζο αναφέρθηκαν στα πρόσφατα γεγονότα στην τουρκία και μετέφεραν στον πρωθυπουργό ερντογκάν με σαφήνεια και συνέπεια τις ανησυχίες της ευρωπαϊκής ένωσης σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της διάκρισης των εξουσιών την ανεξαρτησία και την αμεροληψία της δικαστικής εξουσίας καθώς και την ανάγκη για την ύπαρξη μιας λειτουργικής δικαστικής αστυνομίας. στις συναντήσεις υπογραμμίστηκε ότι η τουρκία ως υποψήφια χώρα έχει δεσμευτεί να εκπληρώσει τα πολιτικά κριτήρια για την ένταξη και ότι είναι σημαντικό να μην σημειώνεται οπισθοδρόμηση και να διασφαλίζεται ότι η δικαστική εξουσία είναι σε θέση να λειτουργήσει χωρίς διακρίσεις και προτιμήσεις κατά τρόπο διαφανή και αμερόληπτο. αναμένουμε συνεπώς από την τουρκία να καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσει ότι πληρεί απολύτω τα κριτήρια της Κοπεχάγης. η εκπλήρωση των κριτηρίων αυτών πέραν του ότι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για αυτή καθεαυτή τη διαδικασία ένταξης είναι προς όφελος της τουρκίας και θα ικανοποιήσει τις θεμητές προσδοκίες των πολιτών της θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σύντομα στι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία σε άλλου τομεί. η ευρωπαϊκή ένωση χαιρετίζει την υπογραφή πέρσι της συμφωνία επανεισδοχή και αναμένει την ταχεία κύρωσή της και την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της εναντί όλων των κρατών μελών. η πρόοδο στο διάλογο για την απελευθέρωση των θεωρήσεων θα βασίζεται στι επιδόσει τη Τουρκία και θα εξαρτάται από την αποτελεσματική και στενή υλοποίηση έναντι της ευρωπαϊκής ένωσης και των κρατών μελών των προαπαιτουμένων περιλαμβάνονται στο σχετικό οδικό χάρτη όπως αυτός συμφωνήθηκε από το συμβούλιο. δεδομένου ότι η τουρκία είναι μία από τις κομβικές χώρες διέλευσης της παράνομης μετανάστευσης προς την ευρωπαϊκή ένωση η ορθή εφαρμογή των υφισταμένων διμερών συμφωνιών επανεισδοχής καθώς και των σχετικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σε ανάλογες συμφωνίες παραμένει προτεραιότητα στο πλαίσιο αυτό η υιοθέτηση του νόμου για τους αλλοδαπούς και τη διεθνή προστασία αποτελεί σημαντική πρόοδο στο πεδίο της μετανάστευσης και του ασύλου. αξιότιμα μέλη βάσει του διαπραγματευτικού πλαισίου και των προηγούμενων συμπερασμάτων ευρωπαϊκών συμβουλίων η τουρκία οφείλει να δεσμευθεί ανεπιφύλακτα ως προς την τήρηση των σχέσεων καλής γειτονίας και την ειρηνική επίλυση των διαφορών σύμφωνα με το χάρτη των ηνωμένων στο πλαίσιο αυτό η ευρωπαϊκή ένωση έχει εκφράσει σοβαρές ανησυχίες και έχει προτρέψει την τουρκία να αποφύγει κάθε είδους απειλή ή ενέργεια στρεφόμενη κατά κράτους μέλους καθώς και οποιαδήποτε πηγή έντασης ή ενέργειας που θα μπορούσαν να βλάψουν τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρηνική επίλυση των διαφορών. επιπλέον η ευρωπαϊκή ένωση έχει τονίσει τη σημασία του σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη σύναψη διμερών συμφωνιών καθώς και την έρευνα και αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών τους βάσει του κεκτημένου της ευρωπαϊκής ένωσης και του διεθνούς δικαίου συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης για το δίκαιο της θαλάσσης. το συμβούλιο έχει επίσης υπογραμμίσει την ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών μελών επί των χωρικών τους υδάτων. σημειώνουμε με βαθιά λύπη ότι η τουρκία παρά τις υποδείξεις συνεχίζει να αρνείται να εκπληρώσει την υποχρέωση πλήρου και άνευ διακρίσεων εφαρμογή του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία σύνδεση έναντι όλων των κρατών μελών. τούτο θα μπορούσε να προσδώσει μια σημαντική όθηση στην διαπραγματευτική διαδικασία. τέλος σαν περισσότερο θετική αναφορά χαιρετίζουμε με ικανοποίηση την επανέναρξη των συνομιλιών με στόχο μια δίκαιη συνολική και βιώσιμη διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος στο πλαίσιο των ηνωμένων εθνών σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του συμβουλίου ασφαλείας και βάσει των αρχών στις οποίες εδράζεται η ένωση. αναμένουμε από την τουρκία να υποστηρίξει ενεργά τις ενεξελίξει διαπραγματεύσεις. η δέσμευση και η συνεισφορά της με συγκεκριμένες ενέργειες σε αυτή τη συνολική διευθέτηση είναι ζωτική σημασία. ευχαριστώ για την προσοχή σας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, χαίρομαι πολύ που σας βλέπω εδώ πέρα, κύριε και κύριοι βουλευτές. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την ε, κυρία Ομνρόιτεν για την ε, συνεισφορά της ε, και το υψηλό επίπεδο του έργου της. της. και για την συνεργασία που είχαμε τα τελευταία 7 χρόνια, αγαπητή μου κυρία. Οι σχέσεις ε, με την Τουρκία βασίζονται σε κάποια στρατηγικά θεμέλια. Οπωσδήποτε η διαδικασία η ενταξιακή είναι η βασική, αλλά και άλλοι παράγοντες έχουν αυξανόμενη σημασία. Οπωσδήποτε ο διάλογος και η συνεργασία στην εξωτερική πολιτική, οι εμπορικές μας σχέσεις, η συνεργασία μας για την κινητικότητα και τη μετανάστευση και ο διάλογος στα ζητήματα ενέργειας. Αυτές είναι πτυχές που καθιστούν την Τουρκία μια ιδιαίτερη χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τελευταίο έτος είχαμε θετικές εξελίξεις, αλλά και λόγια Σταθετικά Στα θετικά ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις στο κεφάλαιο περιφερειακής πολιτικής, το πρώτο κεφάλαιο που ανοίγει εδώ και τρία χρόνια. Υπογράψαμε τη Συμφωνία Επανεισδοχής και ξεκίνησε ο διάλογος απελευθέρωσης των θεωρήσεων. Επίσης ξεκίνησε η αξιολόγηση της Ελληνικής Ένωσης για να αξιολογήσουμε τα θετικά και αρνητικά σημεία που έχει για να επωφεληθούμε ακόμα περισσότερο από τις εμπορικές σχέσεις. Αντιλαμβάνομαι πως η έκθεση της Παγκόσμια Τράπεζας θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή ΙΝΤΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 20 Μαρτίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία συνεχίζουν να έχουν έναν εντατικό διάλογο σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Τέλος, έπαιξε σημαντικό ρόλο η Τουρκία στην επανάληψη των συνομιλιών στην Κύπρο. Δυστυχώς, όπως είπα, είχαμε και λόγους ανησυχίας. Αφορούν κυρίως την αντίδραση της ε, κυβέρνησης ε, στις κατηγορίες περί διαφθοράς, ειδικά όσον αφορά την ε, νομοθεσία για την λειτουργία της δικαιοσύνης και την ελευθερία έκφρασης. Εξέφρασα δημοσίως και απευθείας με τους Τούρκους ομολόγους μου τις ανησυχίες μου. Συνομίλησα μεταξύ άλλων με τον κύριο Ταβουτόγλου και τον Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και βεβαίως και στην έκθεση πρόοδου του Οκτωβρίου θα αναφερθούμε σε αυτές τις εξελίξεις να συνεχίσω και να εμβαθύνω την ε, εμπλοκή μας ε, με τρόπο αποφασιστικό και ειλικρινή με την Τουρκία με βάση το κράτος δικαίου. Αλλά επιπλέον πρέπει να αλλάξει ο τρόπος συνεργασίας για να διασφαλίσουμε πως οι εξελίξει στου διάφορου τομεί πολιτική πηγαίνουν προ τη σωστή κατεύθυνση. Παραδείγματο χάρη πρέπει να συνεργαστούμε στενότερα πριν συνταχθεί η ε, νομοθεσία. Η Κομισιόν θα έρθει σε επαφή με τους ε, ομολόγου μας τι επόμενε εβδομάδες για να υπάρχει μια κοινή αντίληψη επί των αρχών τη συνεργασία μα. Μόνο έτσι θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει παράγων μεταρρυθμίσεων στην ε, Τουρκία και να στηρίξει όσους ζητάνε περισσότερη ευθερία και δημοκρατία στη χώρα αυτή. Εν τω μεταξύ θα συνεχίσω να παροτρύνω το Συμβούλιο να διατυπώσει επιτέλους ε, έναν οδικό χάρτη ή αν θέλετε κάποια συγκριτικά στοιχεία του κεφαλαίου 23 των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Αυτό ζήτησε η ίδια η Τουρκία, οπότε ας τους πιστέψουμε και ας ξεκινήσουμε έναν επικοδομητικό διάλογο για να έχουμε αποτελέσματα στα κρίσιμα αυτά ζητήματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε, και τώρα εκ μέρους του ΕΛ και κυρία Όμιν Ρόιτεν. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους προλαλήσαντες ε, για τα καλά τους λόγια, αλλά βεβαίω ήταν μια συλλογική προσπάθεια με τους συναδέλφους και πάντα ε, ζητούσαμε έναν ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο με την Τουρκία, ο οποίος θα είναι και θα βασίζεται και στην κριτική, αλλά και στην δικαιοσύνη. Και ελπίζω πως ε, πράγματι ε, να επέτυχα ένα θετικό αποτέλεσμα την ε, τελευταία φορά που είμαι εισηγήτρια επί του θέματος αυτού. Κύριε Πρόεδρε, είναι σημαντική η καλή σχέση με την Τουρκία γιατί είναι ένα στρατηγικό εταίρο. Ένα στρατηγικό εταίρο σε μια περιοχή η οποία έχει πάρα πολλέ αναταραχέ. Κύριε Πρόεδρε, το 2005 δεσμεύτηκε για μεταρρυθμίσει η Τουρκία. Τι μεταρρυθμίσει δεν πρέπει να τι κάνει για εμά, αλλά για του Τούρκου πολίτε και έλαβαν χώρα μεταρρυθμίσεις τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά τώρα ανησυχώ, όπως και ο κύριος Επίτροπος και ο κύριος Υπουργός. Ας ξεκινήσουμε τα γεγονότα του Πάρκου Γεζή. τα οποία ξεκίνησαν βεβαίως από τον θάνατο ενός ε, διαδηλωτή, από ένα δακρυγόνο και εδώ πέρα οφείλω να εκφράσω και τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του. Αλλά δεν έχουμε μόνο αυτά τα γεγονότα, αλλά και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις μετά τις 17 ε, Δεκεμβρίου και βεβαίως οπωσδήποτε ασκούμε κριτική στην εκθεσή μας γιατί κυρία Πρόεδρε αυτό το οποίο έχουμε εμείς ως βάση και αυτό είναι μια δέσμευση της Τουρκίας απέναντι μας, απέναντι μας είναι πως θέλουμε ένα κράτος δικαίου και όταν μιλάμε για κράτος δικαίου, εννοείται πως θα υπάρχει μια ανεξάρτητη και αμερόληπτη δικαιοσύνη και δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Κυρία Πρόεδρε, η προστασία της δικαιοσύνης, η προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών, η προστασία της ελευθερίας γνώμης, κυρία Πρόεδρε, αυτά διακυβεύονται αυτή τη στιγμή, γιατί η Τουρκία από ό,τι φαίνεται δείχνει μια ε, εικόνα σεβασμού κάποιων τέτοιων θέσεων. Έγιναν υποτίθεται τον Δεκέμβριο κάποιες σχετικές μεταρρυθμίσεις, αλλά από ό,τι φαίνεται τώρα υπάρχει μια οπισθοδρόμηση. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι πραγματικά ένας πραγματικός επικοδομητικός διάλογος με την Τουρκία και όχι μόνο για την νομοθεσία η οποία έχει ήδη περάσει αλλά και για το μέλλον όπως είπε ο κύριος Επίτροπος. Αυτές είναι νομίζω οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες θα ωφελήσουν και τους Τούρκους πολίτες. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Όμεν Ρόιτεν για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες ο κύριος Όμπιελ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ καταρχήν ως σκιώδης στην έκθεση αυτή θέλω να πω ότι είμαι ικανοποιημένος ε, για την διαδικασία των διαπραγματεύσεων που έλαβε χώρα. Νομίζω ότι είναι ισορροπημένη η έκθεση θετική γιατί αναφέρεται και στις δικές μας επιθυμίες για τη μελλοντική εξέλιξη της Τουρκίας όσο και στις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Δεν θα μπορούσα όμως φυσικά να εκφράσω την ίδια ικανοποίηση την ε, στιγμή της αξιολόγησης της κατάστασης στη χώρα. Έχει περάσει ένας χρόνος ε, από την έκθεση αυτή και δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε αυτό το έτος ε, θετικά. Είδαμε ε, ότι καταστάλθηκαν πάρα πολύ βίαιοι διαδηλώσεις στο πάρκο Γκεζή. Σήμερα μάθαμε ότι πέθανε ο Μουρκενίν Κυρεμπάκ, ο έφηβος που βρισκόταν εννέα μήνες σε γωνία και νομίζω ότι πρέπει να δηλώσουμε τη βούλησή μας να μην επαναληφθούν τις καταστάσεις στη χώρα. Είδαμε και δύσκολες καταστάσεις σε ό,τι αφορά στην κυβέρνηση με την απομάκρυνση διαφορών υπουργών, με το ξέσπασμα σκανδάλων, με τη συνέχιση προβλημάτων που αφορούν ε, τους δημοσιογράφους και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και γενικά ένα πανόραμα βεβαιότητας ενώπιον ενός μέλλοντος που βραχυπρόθεσμα θα είναι αποφασιστικό. Δηλαδή, τι θα συμβεί τους επόμενους ε, μήνες ε, στις ε, δημοτικές εκλογές και στις προεδρικές εκλογές θα είναι καθοριστικά. Εγώ δυστυχώς δεν είμαι σε θέση να κάνω μία πρόβλεψη τώρα σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι ε, θα πρέπει να δηλώσουμε εκ νέου τις επιθυμίες μας και τις δεσμεύσεις μας ε, και να εκφράσουμε με ειλικρίνεια επικρίσεις επί των γεγονότων είναι το καλύτερο που μπορεί να αναμένουμε από μια έκθεση αυτού του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να απευθύνω κλίση σε όλους σας να σέβεστε το χρόνο αγόρευσης ο κύριος ε, Λάμπστορφ εκ μέρους των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, η Τουρκία είναι ένα σημαντικός γειτόνας, μια μεγάλη, περήφανη χώρα. Έχουμε πολλούς Τουρκούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε όλη αυτή την συζήτηση για εμάς τους φιλελεύθερους δεν έπαιξε ποτέ ρόλο το ζήτημα της ε, θρησκείας και θα ήθελα να ευχαριστήσω την συνάδελφο την κυρία Μοντρότην ε, για το ότι η όλη συζήτηση έμεινε σε πολιτικά πλαίσια. Αυτό το οποίο παίζει ρόλο για μας είναι οι ελευθερίες και οι ελευθερίες είναι αυτές οι οποίες απειλούνται στην Τουρκία. Η ελευθερία του τύπου. Είναι πιο πολλοί δημοσιογράφοι φυλακισμένοι στην Τουρκία από ότι στην Κίνα ή στο Ιράν. Στο διαδίκτυο απειλεί ο Πρωθυπουργό να κλείσει το Facebook ή το Twitter, γιατί εκεί πέρα ε, διακινούνται πράγματα που δεν του αρέσουν. Εντάξει, σα φαίνεται τρέλα, αλλά είχε ήδη κόψει μία φορά το YouTube. Αν δούμε το πώς περιορίζεται η κοινωνία των πολιτών από όλο και περισσότερες ε, θρησκευτικές διατάξεις που εφαρμόζονται και πρέπει ο κόσμος να προσαρμόσει την ε, προσωπική του ζωή. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης των δικαστών να μπορούν να κρίνουν το τι ισχύει ε, ή όχι. Και επίσης, από ό,τι φαίνεται, αποκαλύφθηκαν εκατοντάδες ε, περιπτώσεις, ε, ανακάλυψε τώρα η κυβέρνηση, στις οποίες δεν είχε συμπεριφερθεί σωστά η κυβέρνηση και αυτό έγινε μόλις τράφηκε κατά της ίδιας της κυβέρνησης για περιπτώσεις διαφθοράς. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε, όπως είπαμε, αυτή τη μεγάλη σημαντική χώρα στον τομέα της ε, ενέργειας και σε άλλους τομείς. Κάνει πολλά πράγματα η Τουρκία για τους Σύρους πρόσφυγες. Αλλά η σχέση αυτή παραδόξως επιδεινώνεται αντί να ε, βελτιωθεί. Θεωρούμε πως θα πρέπει να ανασταλούν λοιπόν οι συνομιλίες μέχρι να μπορέσει τουλάχιστον η, Τουρκία να σεβαστεί την εξαρτησία της δικαιοσύνης και των πολιτών της. Σας ευχαριστώ. Ο Κόμις του θα ήθελε να σας κάνει μια ερώτηση. Την δέχεστε? Ναι, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ που δέχεστε την ερώτηση. Κύριε Λάμσδοφ, αναφέρατε τη λέξη ελευθερίες στην ομιλία σας. Η Τουρκία θα πρέπει να έχει την ελεύθερη διακίνηση των πολιτών της. Ποια είναι η εκτίμησή σας για τον αριθμό των Τούρκων πολιτών που θα μεταναστεύσουν από την Τουρκία στην Βόρεια Ευρώπη, συγκεκριμένα στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και για να σας βοηθήσω, υπολογίζεται πως ο πληθυσμός της Τουρκίας το 2025 θα είναι 90 εκατομμύρια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Σας έχω άσχημα νέα. Δεν έφερα σήμερα την κρυστάλλινη μπάλα μου εδώ πέρα. Δεν μπορώ να σας πω νούμερα για το οι Τούρκοι θα έχουν το 2025 την ε, ανάγκη να μεταναστεύσουν στη Βόρεια Ευρώπη. Δεν το ξέρω. Αυτό το οποίο μπορούμε όμως να κάνουμε πρακτικά είναι να διευκολύνουμε τις συνθήκες ταξιδιού για επιχειρηματίες, φοιτητές και λοιπούς. Να σταματήσει αυτή η εξευτελιστική κατάσταση ε, να στέκονται στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα και αλλού ουρές οι Τούρκοι μπροστά στα προξενία μας. Θα πρέπει. Όταν λέω εγώ πως θα πρέπει να σταματήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, αυτό σχετίζεται κυρίως με την κυβέρνηση και δεν έχει ούτε μία σχέση όπως είπα με τους ανθρώπους του οποίους πρέπει να διευκολύνουμε. Ευχαριστώ. Τα τελευταία αυτά γεγονότα καθίσουν ακόμη μια φορά σαφές το πόσο σημαντικό να έχουμε μια αξιόπιστη διαδικασία ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Γιατί εάν δεν απέριπταν εκ των προτέρων τα κράτη-μέλη την ένταξη της Τουρκίας θα είχαμε περισσότερο περιθώριο να πιέσουμε. Εάν δεν ε, εάν είχαμε αντιμετωπίσει τα προβλήματα στα ανθρώπινα δικαιώματα, στα θεμελιώδη δικαιώματα κτλ. δεν θα τα είχαμε τώρα μπροστά μας στην δικαιοσύνη. Αλλά αντί να είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχουμε αρχίσει να εξάγουμε τα δικά μας προβλήματα στην Τουρκία, όπως κάνουμε τώρα με τη Συμφωνία Επανεισδοχής. Όλοι γνωρίζουμε πως δεν θα γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των μεταναστών στην Τουρκία, οπότε δεν πρέπει να έχουμε μια τέτοια συμφωνία. Συμφωνούμε πως η απελευθέρωση της βίζας είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο. Ναι, έχουν γίνει σημαντικές ε, δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις τα προηγούμενα χρόνια, αλλά επισκιάζονται από δηλώσεις για την ελευθερία του διαδικτύου και με την βία κατά των διαδηλωτών στο Πάρκο Γκεζί. Και εγώ θα ήθελα να ε, υπενθυμίσω εδώ πέρα τον 17χρονο Μπερκίνερ ο οποίος πέθανε από δακρυγόνα. Επίσης ανησυχώ από τις ε, επιθέσεις στα κόμματα του Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος ε, και ελπίζω να μην σημαίνει αυτό πως δεν θα είναι ειρηνικές εκλογές και οπωσδήποτε οποιαδήποτε πρόοδος επισκιάζεται από το σκάνδαλο αυτό το οποίο μπορώ να ερμηνεύσω μόνο ως απειλή προ την δικαιοσύνη. Αλλά και πάλι ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να είναι πολύ ισχυρότερο εάν είχαμε μια σαφή δέσμευση για θετικό αποτέλεσμα τη συνταξιακή προοπτική. Θα είχαμε πολλά περισσότερα για να πιέσουμε, αν δεχόμασταν πω ναι, θα δεχτούμε την Τουρκία εάν εκπληρώσει τα κριτήρια τη Κοπενχάγη. Αυτό είναι το μόνο το οποίο μετράει και τα κράτη-μέλη πρέπει επιτέλου να είναι σαφή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ομάδα ECR, ο κύριος Βαν Όρδεν, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με τις δημοτικές εκλογές, τα τέλη του μήνα και τις προεδρικές εκλογές αργότερα, ε, φέτος και δεδομένης της ε, κρίσης ε, σε όλη την περιοχή είναι ζωτικό για την Τουρκία και για τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να ρωτήσουμε τι μηνύματα θέλουμε να δώσουμε. Καταρχήν θέλω να πω ότι πολλοί από εμά θέλουν να δουν μεγάλες αλλαγές στην φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτής καθ' αυτής ιδίως. Θέλουμε να μην έχουμε πλέον αιμονή με την πολιτική ολοκλήρωση. Οι πολίτες μας αντίθετα θέλουν να επικεντρωθούν στην οικονομική ανάπτυξη και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του ενσυχεί το θέμα της ελεύθερης κυκλοφορίας ε, και σε αυτούς τους ασταθείς καιρούς προτιμούν την εγγύηση του ΝΑΤΟΚ παρά ε, την ε, μη σοβαρή πολιτική άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, ε, είναι πολύ προς το συμφέρον μας να βάλουμε τα δυνατά μας για να διασφαλίσουμε ότι η Τουρκία συνεχίζει ως ε, μία ε, σταθερή, ελεύθερη αγορά, λαϊκή δημοκρατία και σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Τώρα, η Ευρωπαϊκή, πώς, για πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αποτελεί μία απλώς αγορά για την Τουρκία, αυτό πρέπει να το δούμε και ε, πρέπει να δούμε πόσο οι πολίτες μας είναι διατεθειμένοι να δεχτούν την Τουρκία και με μία μακρά περίοδο μετάβαση. Σας ε, στείλουμε θετικά μηνύματα στην Τουρκία, Σας ανοίξουμε το κεφαλαίο για την ενέργεια, ας δώσουμε νέα όφηση στις διαπραγματεύσεις, Σας αυξήσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσφυγες, στις διασυνορικές περιοχές και ας επικεντρωθούμε στην επανένωση της Κύπρου, αναγνωρίζοντας ότι αυτό είναι ένα θέμα με δύο όψεις που θα βοηθηθεί με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη και από τους Έλληνες και τους Τούρκους. Και ελπίζω ότι η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου θα μπορούσε να συνεισφέρει περισσότερο σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα. Ευχαριστώ. Uh, there is a blue card. Υπάρχει μια μπλε κάρτα για σας. Τζέφρε, συμφωνείτε με την εξή. πρόταση να γίνει πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι το πιο ευέλικτο όπου παραδείγματο χάρη το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει μια πιο χαλαρή σύνδεση στις ε, χώρες οι οποίες επιμένουν σε αυτή την πολιτική ολοκλήρωση που σας ενοχλεί και μετά η Τουρκία θα έχει τον ίδιο βαθμό σύνδεσης με το Ηνωμένο Βασίλειο σε αυτή την Ευρώπη των δύο ταχυτήτων νομίζω πως θα ήμασταν όλοι χαρούμενοι αν η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πιο χαλαρά συνδεδεμένοι, οι υπόλοιποι να μπορούν να προχωρήσουν. Θα σας ικανοποιούσε κάτι τέτοιο. Χωρίς μικρόφωνο. Έχετε απολύτως δίκιο. Θα ήταν θετικό αυτό. Κάτι τέτοιο θα θέλαμε στη χώρα μας. Δεν μου αρέσει βεβαίω αυτό το οποίο είπατε για δύο ταχύτητε, γιατί το πιο γρήγορο ακούγεται πιο ωραίο. Εγώ θα το έλεγα μια Ευρώπη με πολλά κέντρα ή με αλληλεπικαλυπτόμενου ε, κύκλου ή αλακάρτ. Οπωσδήποτε με το Ηνωμένο Βασίλειο στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά χωρίς να εμπλέκεται σε πολλούς τομείς όπου εσείς θέλετε περισσότερη ολοκλήρωση. Και νομίζω με αυτή τη βάση θα είναι και πολύ πιο εύκολο για την Τουρκία να γίνει μέλος. Ευχαριστώ για την ομάδα ΚΟΕ. Ο κύριος Χατζηγεωργίου για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν πρέπει να πω ότι είναι πάντα μια ωραία πρόκληση να μιλά κανείς <clears throat> μετά τον συνάδελφο τον κύριο Βαν Όρντεν, τον καλύτερο ίσως πρεσβευτή της Τουρκίας στο Ευρωκοινοβούλιο Εμεί εκφράζουμε την πεποίθηση ότι τα πράγματα που τρέχουν σήμερα στην τουρκία πρέπει να μα απασχολούν θετικά να μας απασχολούν γιατί μας ενδιαφέρει οι αντιπαραθέσει που ε, συμβαίνουν σήμερα στην τουρκία να μην σπρώξουν την τουρκική κοινωνία προ τα πίσω και πω το περιεχόμενο των οποιοδήποτε μεταρρυθμίσεων σήμερα στην τουρκία δεν θα ξεπαστρέψει τους αδύνατου και δεν θα οδηγήσει τους πολίτε τη χώρα σε κοινωνικό και εργασιακό μεσαίωνα με αυτά υπόψη ο δικό μα ρόλο πρέπει να είναι θετικό απέναντι στην τουρκία. αυτό όμω προτάσσει πρωτίστω την αντικειμενική αντίκριση των δεδομένων αυτή τη χώρα και των δεσμεύσεών τη. συγχαίρουμε την εισηγήτρια για την προσπάθειά τη και επισημαίνουμε πω υπάρχουν περιθώρια βελτίωση. ενδεικτικά για μα είναι παράλογο να ασκούνται πιέσει για το άνοιγμα των κεφαλαίων 15, 23 και 24 όταν η τουρκία επιμένει σε μη υλοποίηση των σχέσεών της ομαλοποίηση των σχέσεών της με την κυπριακή δημοκρατία αρνούμενη να υλοποιήσει το πρωτόκολλο το οποίο έχει ήδη υπογράψει και αρνούμενη να αναγνωρίσει ή να της επιτρέψει να εφαρμόσει συναφώς τα κυριαρχικά της δικαιώματα. η εφαρμογή του δικαίου του ισχυρού είναι που έφερε την τουρκία στην κύπρο και εμείς είμαστε ενάντια στο δίκαιο του ισχυρού. πρέπει να πω εδώ ότι εμείς στηρίζουμε την επανέναρξη των συνομιλιών στην κύπρο και ελπίζουμε να καταλήξουν θέλουμε να καταλήξουν γιατί εμεί πρωτίστω είμαστε αυτοί που υποφέρουμε από την διέρεση και την κατοχή και αναμένουμε ω εκ τούτου από την ευρωπαϊκή ένωση και από ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα να σταθεί αλληλέγγυα στον αγώνα για τερματισμό του διχοτομικού status quo για μια λύση διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία που να σέβεται το διεθνέ δίκαιο να διασφαλίζει το αδιέρετο τη πατρίδα και του λαού μα και να αποστρατιωτικοποιεί την κύπρο. δέκα δευτερόλεπτα κυρία πρόεδρε να πιέσει την τουρκία να επιτρέψει την εφαρμογή οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνη που να μην αφήνουν υπονοούμενα αναβάθμιση του ψευδοκράτου όπω το απευθεία συμπόριο. και υπενθυμίζω την πρόταση για παράλληλη εφαρμογή του ψηφίσματο 550 του Συμβουλίου Ασφαλεία για την Αμόχωστο με τη λειτουργία του λιμανιού και τον τερματισμό του παράνομου επικισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ομάδα EFD, ο κύριος Σαλαβράκος, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαιρετίζω και εγώ με τη σειρά μου την έκθεση της κυρίας Όιμεν Ρόιτεν, η οποία συμπληρώνει προηγούμενες εκθέσεις της και παρουσιάζει κατά το δυνατόν την κατάσταση που υπάρχει στη χώρα αυτή, αποτελώντας με τις προηγούμενες εκθέσεις της ένα ενιαίο όλων, καθό μέρος δεν τις αναιρεί ρητά αναμφισβήτητα η τουρκία είναι μια σημαντική οικονομική δύναμη και μια χώρα με αυξημένο γεωπολιτικό ρόλο στην περιοχή της μέσης ανατολής. ωστόσο η χώρα αυτή απέχει πάρα πολύ από τα ευρωπαϊκά πρότυπα δημοκρατικών αρχών και αξιών. όπως πολύ σωστά επισημαίνει η εισηγήτρια μέσα από την έκθεσή της η εσωτερική κατάσταση στην τουρκία είναι ανησυχητική χαρακτηρίζεται από σκάνδαλα διαφθορά υιοθέτηση νόμων που θέτουν υπό αμφισβήτηση τη συνταγματική διάκριση των εξουσιών και τα θεμελιώδη δικαιώματα όπω παράδειγμα ο πρόσφατο νόμος για τη διαδικτυακή λογοκρισία και την αύξηση των εξουσιών τη Εθνική Μυστική υπηρεσίας. η τουρκία αρνείται πεισματικά να υπογράψει διεθνεί συμφωνίε, όπω την unclos δεν τηρεί τα συμφωνημένα με την ευρωπαϊκή ένωση δεν έχει εφαρμόσει για όγδοη συνεχή χρονιά τις διατάξεις που απορρέουν από τη συμφωνία σύνδεσης ευρωπαϊκής ένωσης τουρκίας και το πρόσθετο πρωτόκολλό της δεν αναγνωρίζει κράτος μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης εξακολουθεί η απειλή του κάζους μπέλικα κατά της ελλάδος συνεχίζονται οι παραβιάσεις των ελληνικών χωρικών υδάτων και δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα κρατών μελών της ένωσης. εξώνυχος τον λέοντα. επιπρόσθετα σημειώνω ότι η ευρωπαϊκή ένωση στα πλαίσια της προενταξιακής βοήθειας έδωσε 900 εκατομμύρια για το 2013 στην Τουρκία. Θα πρέπει επιτέλους να επανεξεταστεί γενικότερα η πορεία της Ένωσης και να συγκεντρωθούμε στα σημαντικά προβλήματα που αφορούν τους πολίτες της Ένωσης. Αυτό ζητάμε από εμάς οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ο λόγος της διπλωματίας ενίοτε ωρεοποιεί καταστάσεις και παραβλέπει γεγονότα την επέλευση όμως των οποίων δεν αποτρέπει. χρειάζεται καθαρός λόγος προς την τουρκία. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σα παρακαλώ να σέβεστε το χρόνο αγόρευση, Ένα μισή λεπτό κύριε Λίζεκ. Όχι, με συγχωρείτε. Στράσεν για του μη Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως πάντα βλέπουμε να προκαλεί τα πάθη η Τουρκία. Το μοναδικό συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε είναι πως η Τουρκία δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα, δεν μπορεί να γίνει και δεν θα προσχωρήσει ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από ό,τι φαίνεται πάνε πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα στην Τουρκία για τον Ισλαμιστή Ερντογάν. Βλέπουμε αφενός την καταστολή με την αστυνομία, την υπονόμευση του κράτους δικαίου και το περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης. Δεν είναι δυνατόν πλέον μετά από όλα αυτά να πούν κάτι διαφορετικό η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε από το Συμβούλιο να αναστείλει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Το ερώτημα είναι γιατί δεν το κάνει αυτό η Κομισιόν και η απάντηση είναι πως η Κομισιόν θέλει οπωσδήποτε να προωθήσει την ένταξη της Τουρκίας. Όμως το κόμμα το κόμμα της ελευθερίας έχει αντίθετη άποψη. Το Ισλαμιστικό κατασταλτικό κράτος Τουρκίας δεν πρέπει ποτέ να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να το επιτύχουμε αυτό, σας καλώ να ψηφίσετε στις ευρωεκλογέ το ΠΒΔ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ. Κύριε Επίτροπε. Εδώ μιλώ ως Ευρωπαίος αλλά και ως Πολωνός πολίτης. Γιατί αναφέρω το τι είμαι Πολωνός ε, φέτος. Η Πολωνία και η Τουρκία γιορτάζουν ε, την ε, εξεκουσιστή επαιτίο τη σύνοψη διπλωματικών σχέσεων. Οι σχέσει της Πολωνίας με την Τουρκία ήταν πάντοτε πολύ καλές και η Τουρκία ήταν η μόνη χώρα που δεν αναγνώρισε τη διχοτόμηση της Πολωνίας το 18ο αιώνα και κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο προστάτευσε την πολωνική πρεσβεία από τους Ναζί. Έχουμε λοιπόν ε, καλή ιστορική συνεργασία και εδώ θα ήθελα να παροτρύνω την Τουρκία να αναλάβει τις απαραίτητες δράσεις προκειμένου να εκπληρώσει όλες τις απαιτήσεις που έχει ως υποψήφια προσέντεξη χώρα η Τουρκία, όπως και όλες ε, οι υπόλοιπες χώρες, πρέπει να εκπληρώσει τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Θα πρέπει να δείξει ότι σέβεται τις ευρωπαϊκές μας αξίες, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει να δείξει ότι καταπολεμά τη διαφθορά. Θα πρέπει να επικεντρωθεί σε όλες τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να επιταχύνει τη διαδικασία της προσχώρησης, όμως ε, ιδίως στη μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χαουίτ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε και εγώ θα αναφερθώ στον Θάν Μπερκίν Ελφάν ο οποίος είχε βγει να αγοράσει ψωμί και τον σκότωσε ένα δακρυγόνο της αστυνομίας και πέθανε σήμερα στα 15 του καθώς ήταν σε κόμμα τόσο καιρό και οι διαμαρτυρίες όπως αναφέρει η Εθνής Αμνηστή αποτελούν μέρος των συνεχών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Τουρκία, από ό,τι φαίνεται, καταστέλει την αντιπολίτευση. Πάνω από 50 δημόσιοι υπάλληλοι συνελήφθησαν τον προηγούμενο μήνα γιατί ανήκαν σε ένα συγκεκριμένο συνδικάτο, το οποίο, κατά το οποίο βέβαια καταδικάζει και η Διεθνής Ομοσπονδία Συνδικάτων, όπως επίσης και τη χρήση της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας για το θέμα αυτό. Επίσης υπάρχει ολική υπάρχει μπλοκάρισμα της πρόσβασης στο YouTube και στο Facebook που παραβιάζει την ελευθερία έκφρασης και υπάρχει και ο νέος νόμος για το Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελίων ο οποίος παραβιάζει την διάκριση των εξουσιών και σύμφωνα με το Human Rights Watch από ό,τι φαίνεται η πολιτική θα έχει μεγαλύτερη εξουσία επί της δικαιοσύνης. Η Τουρκία μπορεί να τα πάει καλύτερα από έτσι. Σας ευχαριστώ κύριε Σντάφ για 1,5 λεπτό. Η κρίση αυτή Ε, που έχει ξεσπάσει στο τουρκικό κράτος ε, ενισχύεται συνέχεια ε, και αυτό κυρίως του ρήγματος μεταξύ του κυρίου Γκιουλέν και του κυρίου Ερντοάν. Νομίζω ότι για να φανούμε αξιόπιστοι η έκθεση του κοινοβουλίου μας θα πρέπει να αναφέρεται σε αυτή την πτυχή ε, που χρωματίζει την κρίση. Ο κύριος Φούλε αναφέρθηκε σε σοβαρές ανησυχίες. Πρέπει να σας πω εγώ πως λυπάμαι ιδιαίτερα πως οι ανησυχίες αυτές είναι τόσο πλέον σοβαρές όπου η Τουρκία πλέον δεν πληρεί επαρκώς τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Το φθινόπωρο λοιπόν η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η νέα θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να εξετάσουν κατά πόσο αυτές οι ε, μακρόχρονες και ε, μακροσκελείς ε, ενταξιακές διαπραγματεύσεις είναι βιώσιμες. Και θα πρέπει να σκεφτούμε εάν ίσως κάποια εναλλακτική σχέση η μορφή ε, ένταξης η οποία δεν θα είναι ε, με την ιδιότητα του πλήρους μέλους θα ήταν ενδεχομένως ε, μια καλύτερη διαφθέτηση προς όφελος και της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Grazie. Onorevole. Ευχαριστώ. Κύριος Μπέλντερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. 18 Απριλίου 2007 ήταν μια μαύρη ημέρα για την προτεσταντική κοινότητα της Τουρκίας γιατί τη μέρα εκείνη πέντε νεαροί Τούρκοι γιόρταζαν το μίσος τους κατά της χριστιανοσύνης δολοφονώντας έναν ιερέα στην Μαλάτια. Και σήμερα η μικρή προτεσταντική κοινότητα της Τουρκίας είναι σοκαρισμένη. Γιατί, από ό,τι φαίνεται, με μια πρόσφατη απόφαση απελευθερώθηκαν οι πέντε δολοφόνοι αυτοί. Αντιλαμβάνεστε πως έχει σοκαριστεί η προτεσταντική κοινότητα της Τουρκίας για το ότι οι εγκληματίες κατά τη διάρκεια της δίκης απειλούσαν ανοιχτά τους χριστιανούς, τους συγγενείς των θυμάτων, τους δικηγόρους τους, τα ΜΜΕ και όποιον έβρισκαν μπροστά τους. Και τώρα απελευθερώνονται. Οι προτεστάντες στην Τουρκία φοβούνται. Έχουν στείλει μια ανοιχτή επιστολή. Φοβούνται για την ζωή τους. Και απευθύνω έκκληση σε εσά. Επίτροπε, να μιλήσετε στις τουρκικές αρχές και να ζητήσουν την ισόβια καταδίκη αυτών των δολοφόνων. Αφέθηκαν ελεύθεροι. Είναι απαράδεκτο να συμβαίνει αυτό σήμερα Και κάτι άλλο. Εξακολουθεί να υπάρχει αντισημιτισμός διαρκής στα τουρκικά μήμια, το οποίο το ανέχονται οι τουρκικές αρχές. Απαράδεκτο για μια χώρα η οποία είναι υποψήφιο μέλος. Δεν έχει ουδεμία σχέση μεταξύ μα και δεν επιτρέπεται να σιωπούμε. Ο Στάντλερ, για ένα λεπτό. Θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ στο θέμα αυτό. Κάποιοι αναφέρθηκαν στον δολοφονημένο Μπέρκιν Ελβαν. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στον Τέλμαν Γκίσκ, Γερμανό δολοφονηθέντα ε, προτεστάντη οι άνθρωποι αυτοί που δολοφονήθηκαν βασανίστηκαν επί ώρες και μετά τους πυροβόλησαν στο λαιμό και κυκλοφορούν ελεύθεροι οι δολοφόνοι. Αυτή την Τουρκία θέλετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγχαρητήρια, τι να σας πω. Την Τουρκία που επιτρέπονται τα πάντα. Έτσι, η κατάσταση επιδεινώθηκε από την τελευταία φορά που συζητήσαμε με τον λεγόμενο νόμο περί δικαιοσύνης, με τον νόμο περί ίντερνετ. Κάθε χρόνο και χειρότερα. Αλλά εσεί επιτρέπετε τα πάντα στην Τουρκία. Αν τα έκανε αυτά η Ρωσία, ξέρετε τι θα γινόταν εδώ μέσα. Με την Τουρκία τίποτα, έτσι δεν παίζει τίποτα ρόλο. Γιατί, γιατί είστε υπό τον ζυγό των στρατηγικών και οικονομικών συμφερόντων. Αυτή είναι η ηθική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πάντα εξαρτώνται από το ποιο κάνει κάτι. Έτσι. Η, Ευρώπη, η Τουρκία δεν ανήκει στην Ευρώπη. Και σας εγγυώμαι πως εάν προσπαθήσετε να την βάλετε θα καταψηφίσουν οι Αυστριακοί στο δημοψήφισμα. Ναι, ευχαριστώ. Ο κύριος μόνο για ένα μισή λεπτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγητρία για την πλήρη έκθεσή της. Είναι πολύπλοκη διαδικασία ένταξης της Τουρκίας Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει οδηγήσει την Τουρκία ε, στο να κάνει μεταρρυθμίσεις και πρέπει να συνεχίσει αυτή την οδό και να μην υπενοχωρήσει σε σχέση με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το κράτος δικαίων, εξαρτία τη δικαιοσύνη. Αυτοί είναι πυλώνες του αρχιτεκτονική ενό ευρωπαϊκού κράτου, Οι αρχέ. Ε, τις Τουρκίες πρέπει να σέβονται πλήρως αυτές τις αρχές, μάλιστα όταν βιώνει η χώρα κρίσιμες στιγμές. Γι' αυτό πρέπει να μελετήσουμε την θετική στάση της εισήγησης της κυρίας Όμων και νομίζω ότι πρέπει να ανοίξετε τα κεφάλαια 23 και 24 σύντομα. Αυτό θα επιτρέψει στην Ένωση να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυ σε αυτά τα τόσο σημαντικά θέματα για τη δομή του κράτους. Από την άλλη, ε, χαίρομαι για την υπογραφή της Συμφωνίας Επανεσδοχής λόγω της γεωγραφικής της θέσης η Τουρκία διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ε, ε, στον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών που έρχονται προς την Ένωση και η πολιτική της για τη χορήγηση θεωρήσεων για τρίτες χώρες θα πρέπει να είναι αντικείμενο στενού συντονισμού με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν γίνεται κάτι τέτοιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια κρίσιμη στιγμή για το θέμα της γειτονίας. Ε, είχαμε ε, την Αραβική Άνοιξη, έχουμε την κατάσταση στην Ουκρανία και τον πόλεμο στη Συρία. Η χώρα, η Τουρκία, θα πρέπει να είναι είναι ένας ε, εταίρος με τον οποίο θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει έναν έντονο διάλογο για τις σχέσεις με τις γειτονικέ χώρες. Ευχαριστώ κυρία Κοπά. Σήμερα στις 7 το πρωί, την ίδια τη μέρα που στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητάμε για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, ένα 15χρονο παιδί, ο Μπερκίν Ελβάναυσε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο στην Κωνσταντινούπολη. Ο Μπερκίν χτυπήθηκε από δακρυγόνο τον Ιούνιο στα γεγονότα του πάρκου Γκεζί εκείνη την ώρα δεν συμμετείχε στη διαδήλωση πήγαινε να αγοράσει ψωμί και από τότε έμεινε 269 μέρες σε κόμμα. Ο θάνατος αυτός είναι ο όγδοος που σχετίζεται με τα γεγονότα του πάρκου Γκεζί και αυτός όπως όλοι οι άλλοι θα μείνει ατιμόρυτος. Η οικογένεια του παιδιού κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προστατεύει τους ενόχους. Δεν υπήρξε όμως καμία αντίδραση. Ας μην ξεχάσουμε εδώ στο Κοινοβούλιο τα γεγονότα του πάρκου Γκεζί τα αιτήματα για περισσότερη δημοκρατία διαφάνεια λογοδοσία δεν έχουν βρει ανταπόκριση. η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνεχίζει να χειροτερεύει και όσο ο κύριος ερντογάν είναι σε αμφισβήτηση λόγω διαφθοράς το κατασταλτικό σύστημα γίνεται όλο και πιο σκληρό. ο σημερινός τραγικός θάνατος ενός μικρού παιδιού μας καλεί όλους να ενώσουμε τη φωνή μας για πραγματική δημοκρατία στην τουρκία και για ένα οριστικό τέλος στην αστυνομική βία στην τουρκία και παντού εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. πολύ. Γεωγραφικά η Τουρκία είναι 97% στην Ασία. Παρ' όλα αυτά η τουρκική κυβέρνηση ακολουθεί μια στάση ε, που την τοποθετεί 100% στη Μέση Ανατολή όταν έχει αντιρρησίες. Όπως και η Κούβα έχει ένα νόμο περιορισμό του διαδικτύου. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να ε, περιορίσει τις δικαιοσύνες των εισαγγελέων και των δικαστών. Είναι πολύ οι φυλακισμένοι δημοσιογράφοι στην Τουρκία και ο κύριος Ερντοάν μας είπε με μεγάλη υπερηφάνεια πως μίλησε για το θέμα αυτό ε, και μας είπε και ο κύριος Φούλε ότι τα είπανε με τον κύριο Εντοάν και με ε, τους Τούρκους. Ξέρετε πως τέτοιου είδους φαινόμενα δεν αρμόζουν σε μια δημοκρατία. Η Τουρκία δεν ακολουθεί τις δυτικές αξίες. Η Τουρκία θα έπρεπε να θεωρείται ως υπερβολικά μεγάλη, υπερβολικά φτωχή, υπερβολικά διαφορετική, υπερβολικά αυταρχική για να γίνει ποτέ μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι πραγματικά απογοητευτικό που η τα κόμματα του συστήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο στηρίζουν την πρόσβαση της χώρας αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει και αυτοί και εσείς να το ξανασκεφτείτε. Ευχαριστώ κύριος Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μα τι πρόοδος, τι πρόοδα μιλάμε αγαπητοί συνάδελφοι. Αναγνωρίζετε τη γενοκτονία των Αρμενίων ή των Βουλγάρων επί πέντε αιώνες στη Βουλγαρία η Τουρκία έχει δώσει κάποιες αποζημιώσεις για τους μετανάστες της Θράκης ε, του 13 έχει απελευθερώσει τους ε, δημοσιογράφους έχει ε, επικυρώσει την συμφωνία πανισδοχής η Τουρκία δεν χρησιμοποίησε αστυνομική δύναμη για να εξαλείψει τις φωνές αντίδρασης. Ε, τι κάνει ο κύριος Ερντοάν, δεν συνεχίζει να κατέχει η Τουρκία κομμάτι της Κύπρου. Πού είναι η θετική εξέλιξη, τι έκανε η Τουρκία για να σταματήσει η βία εναντίον των χριστιανών. Οι διαπραγματεύσεις με την Τουρκία θα πρέπει να διακοπούν αμέσως, όχι στην Τουρκία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, κυρία Γιαννάκου. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ε, άκουσα με προσοχή την Προεδρία καθώς και τον Επίτροπο. Είναι γεγονός ότι η έκθεση αυτή για την κατάσταση στην Τουρκία έχει αρκετά στοιχεία υπέρ της Τουρκίας και θετικά. Εν τω μεταξύ όμως πάρα πολλά από όσα έχουν υποθεί έχουν διαψευστεί από την πραγματικότητα ε, η έλλειψη πολιτικής σταθερότητας και τα σχόλια γύρω από την ηθική κατάσταση σε σχέση με την κυβέρνηση ε, τα επεισόδια που γίνονται κάθε φορά στο πάρκο γκεζί ο θάνατος πολλών ατόμων οι δημοσιογράφοι που είναι στη φυλακή το ζήτημα της δικαιοσύνης γενικότερα οι αμφισβητήσεις που υπάρχουν και ας υποθέσουμε ότι όλα αυτά προέρχονται από αναταραχές που προκαλούνται για διαφόρους λόγους ωστόσο υπάρχουν τα ζητήματα που εξαρτώνται αποκλειστικά από την κυβέρνηση δηλαδή η αναγνώριση του συνόλου της ευρωπαϊκής ένωσης η αναγνώριση του πρωτοκόλλου της άγκυρας δηλαδή η συνέπεια σε σχέση με αυτό που η τουρκία επιδιώκει. υπάρχουν ακόμα ερωτηματικά για το αν η τουρκία θέλει να γίνει μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης. πιστεύω αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει δεν πρέπει να υπάρχουν υποθέτουμε ότι η τουρκία θέλει να γίνει μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης θέλει όμως να γίνει μέλος όπως είναι χωρίς να αλλάξει τίποτα και αυτό είναι ένα μεγάλο πολιτικό ζήτημα το οποίο πρέπει να κριθεί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι με πολιτικούς όρους. βεβαίως η προσπάθεια αυτή προς την ένωση βοηθά την ίδια την τουρκία να βελτιώσει την κατάστασή της έστω και επιφανειακά αλλά επί της ουσίας για το αν θα γίνει μέλος ή όχι της ένωσης τα ερωτηματικά εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν για το αν πραγματικά το θέλει ή το επιδιώκει. Ευχαριστώ. Το λόγο ο κύριος Σοφοκλέους για ένα λεπτό. Η το επιδιωκει για ενα η τουρκια συνεχιζει να φυλακίζει δημοσιογράφους, πνευματικούς ανθρώπους, φημώνει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης καταστέλει βιε κινητοποιήσεις πεθαίνουν άνθρωποι από τις συμπεριφορές του ερντογάν. ο περκίλ δεν είναι στη ζωή. τα σκάνδαλα πλέον δεν είναι είδηση είναι καθημερινότητα. απειλεί την ευρωπαϊκή ένωση ασκεί μια πολιτική αντιευρωπαϊκή δεν σέβεται θεσμούς δεν σέβεται τη διεθνή νόμη τάξη ψηφίσματα του οργανισμού ηνωμένων εθνών δεν αναγνωρίζει την κυπριακή δημοκρατία δεν βοηθά στην επίλυση του κυπριακού προβλήματο. η έκθεση δεν είναι ισορροπημένη. απλά καταγράφει γεγονότα δεν αναδεικνύει τα μεγάλα ανοιχτά προβλήματα και το κυριότερο δεν καταγράφει δραστικές προτάσεις που θα βοηθούν την εκδημοκρατικοποίηση της χώρας και θα ενισχύουν τις προσπάθειες του τουρκικού λαού. είναι η ώρα η ευρώπη να αντιδράσει να μην επιτραπεί να ανοίξει το κεφάλαιο 15, 23 και 24. Επιτέλους Α στείλουμε το μήνυμα ότι η ευρωπαϊκή ένωση έχει φωνή και επιβάλλεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Κουρκουλα, κύριε Πίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, εκατοντάδε χιλιάδε ε, πολίτε από το Ταξίν και τον Κεζί δήλωσαν ότι δεν υπάρχει δημοκρατία στην Τουρκία. Παραβιάστηκαν οι προσωπικέ ελευθερίε, η ελευθερία έκφραση, η ελευθερία του συνεταιρίζεστε. Τα σκάνδαλα και η διαφθορά είναι πανταχού παρόντα. Η κυβέρνηση εμποδίζει την λειτουργία του δικαστικού συστήματος. Έχουμε δει κάποια παραδείγματα όπως η δίκη Εργένεκον. Η Τουρκία παραβιάζει ε, την ακαιρεότητα ε, της Βουλγαρίας χρησιμοποιεί ε, την μειονότητα στη Βουλγαρία για να θέσει σε εφαρμογή νεοοθωμανικές στρατηγικές. Έχει στο στόχαστρο ε, κάποιες περιοχές που πολιτικά και οικονομικά εξαρτώνται από την Τουρκία. Νομίζω ότι αν η Τουρκία δεν προβεί σε βαθιές μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό της και συνταγματικό της σύστημα, δεν έχει θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς ε, θα πρέπει να ασκήσουμε μια καλή πολιτική γειτονία με τη συνεργασία της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Κύπρου. Ευχαριστώ κυρία Θεοχάρους για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Μα ζητήσατε να τους πιστέψουμε αλλά αυτή τη στιγμή στην Τουρκία υπάρχει γενικευμένη εξέγερση. Τα, οι τηλεοράσεις μεταδίδουν τα γεγονότα, οι παρουσιαστές φορούν μαύρα, δεν ξέρω για πόση ώρα ακόμα. Αυτό όσον αφορά το εσωτερικό της Τουρκίας. Όσον αφορά το εξωτερικό, δύο τουρκικά υποβρύχια, η φρεγάτα Ήμβρο και το Μπάρπαρος περιπονούν στις ακτές της Κύπρου, στις δυτικές ακτές της Κύπρου και συνεπώ εγώ δεν μπορώ να του πιστέψω κύριε Επίτροπε. Από την άλλη είχα ενθαρρυνθεί από τη δήλωση του, Ευρωπαίου, του Τούρκου ε, ε, πρέσβη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είπε ότι το Κυπριακό είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην ενταξιακή πορεία τη Τουρκία. Και είχαμε πει ότι ε, κατάλαβαν επιτέλου και αυτοί ότι πρέπει να λυθεί το Κυπριακό. Αλλά κύριε Υπουργέ δεν μα είπατε ότι στην Κύπρο δεν είναι διαφορά μεταξύ γειτονικών κρατών αλλά είναι εισβολή και κατοχή και συνεπώ ω τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται. Ο ταλαιπωρημένος και φοβισμένος Κυπριακό λαός, αγαπητοί συνάδελφοι, επερίμενε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα θέσει του όρους, θα θέσει τις προϋποθέσεις της επίλυσης του κυπριακού προβλήματος που θα ήταν οι βασικές αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως έπραξε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα προχθέ στο μανιφέστο του στο ε, Δουβλίνο. Ανταυτού κύριοι συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος έρχεστε και μας λέτε ένα περίγραμμα λύσης του κυπριακού προβλήματος το οποίο ερμηνεύει ο καθένας όπως θέλει δεν διασφαλίζει τίποτα και δίνουμε άλοθη στην αυθαιρεσία και στην δύναμη της τουρκίας την οικονομική που τόσο πολύ θαυμάζεται να επιβάλλεται ε, στην, ε, στην ε, περιφέρεια. αυτό δεν συνάδει με τις αρχές και αξίες της ευρωπαϊκής ένωσης και καλά κάνετε να το αναθεωρήσετε. η έκθεση είναι εκτός τόπου και χρόνου το ίδιο και η συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Ε, που παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς ε, τα τεκτενόμενα στην Τουρκία άκουσαν αρχικά ότι υπήρχε σοβαρή απειλή για τη δημοκρατία στην Τουρκία όσοι ήταν ε, υπευθυνοί ε, και σχεδίαζαν στρατιωτικό πραξικόπημα έπρεπε να τιμωρηθούν. Τώρα ακούμε ότι όλα αυτά ήταν συνωμοσία. Υποπτήσει στι συναφείς υποθέσεις απελευθερώθηκαν. Φυσικώς καλωσορίζουμε την απελευθέρωση δημοσιογράφων και άλλων που κρατούνταν για χρόνια. Όμως όσοι είναι ύποπτοι για τη δολοφονία μελών Λοιπόν, του Κρατικού Συμβουλίου ε, έχουν επίσης απελευθερωθεί. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Ε, και είναι ασαφές ε, πλέον τι να πιστέψουμε. Η αλήθεια φαίνεται να μετακινείται ανάλογα με το ποια εφημερίδα διαβάζει κανείς και σε μεγάλο βαθμό ο λαός ε, της Τουρκίας ε, χάνει την πίστη του στο κράτος δικαίου και στο ρόλο της δημοκρατίας, δηλαδή στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία θα πρέπει να επανέλθει στο εινοδό των μεταρρυθμίσεων και να λάβει όλα τα μέτρα για να ε, δώσει πίσω στο λαό της Τουρκίας το πιστεύω του στη δικαιοσύνη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τύρια, ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν ε, θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια για την πολύ ισορροπημένη έκθεση. Η Τουρκία είναι μια πολύ σημαντική χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω ε, για μια χώρα όπως η Κροατία. Λόγω της ε, γεωγραφικής της θέσης. Η Τουρκία είναι σημαντικός παίκτης και έχει δείξει κάτι τέτοιο όταν διαδραμάτισε έναν επικοδομητικό ρόλο στην λήξη της ε, σύραξης στη Βοσνία Ριζεγοβίνη και συνεχίζει να παίζει σημαντικό ρόλο, όμως συχνά ακούμε από την τουρκική ηγεσία κάποιες διαφορετικές φωνές και αισθανόμαστε ότι θέλουν να επεκτείνουν το πεδίο επιρροής τους στην πρώην Οθωμανική Αυτοκρατορία στα εδάφη της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ακούσαμε και τι είπε και ο κύριος Ερντογάν, ότι η νίκη του στις εκλογές είναι σημαντική και για την Κωνσταντινούπολη ως και για την Βεριτό και είπε ότι του αφέθηκε ως ε, μέρος της κληρονομιάς ε, του η Βοσνία σε αυτόν. Δεν θέλουμε να ακούμε ε, τέτοια λόγια εμείς μιλάμε εδώ για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Δεν θέλουμε να επιστρέψουμε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Τουρκία πρέπει να δεκτεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα και γι' αυτό καλωσορίζω το γεγονό ότι η Τουρκία καλείται να ευθυγραμμίσει την πολιτική της προ τη Βοσνία Ζεγοβίνη με την πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκρίσμπεχ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. πολύ. Η Τουρκία είναι μία χώρα ε, από τους μεγαλύτερους εταίρους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Είναι μια χώρα που προσπαθεί να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πολλά χρόνια και αυτή τη στιγμή τρέχουν οι ενταξιακέ διαδικασίε. Και όσο συνεχίζονται, μπορούμε να κάνουμε πολλέ αλλαγέ. Γι' αυτό θα ήθελα να τονίσω σήμερα πω για οποιοδήποτε θέμα, όπω τα ε, θεμελιώδη δικαιώματα, τι βασικέ ελευθερίε, πάρα πολλά ακόμα μπορούν να γίνουν. Όμω, χρειαζόμαστε να ξεκαθαρίσουμε. Ε, το ότι έχει σημειωθεί πρόοδος και κυρίως τα θέματα των μειονοτήτων. Δεν μιλώ μόνο εδώ για την κουρδική ε, μειονότητα αλλά και για τους ε, Κούρδους του Ιράκ. Αυτό που με ανησυχεί είναι η ελευθερία έκφρασης, η φυλάκιση δημοσιογράφων και βεβαίως η βία κατά της ανταπολίτευσης. Εάν δεν λυθούν τα ζητήματα αυτά, η Τουρκία δεν θα μπορεί καν να σκέφτεται την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως το ίδιο ισχύει και για ε, το, τη λύση του Κυπριακού. Έχουμε λάβει κάποιες πληροφορίες ε, για προσπάθεια χειραγώγηση του διαδικτύου, για παράδειγμα, στην ε, Τουρκία. Ίσως ο Πρωθυπουργό τελικά να κάνει πίσω. Και νομίζω πως αυτό θα αποτελούσε ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Νομίζω πως πρέπει να συνεχίσουμε το διάλογο με την Τουρκία. Είναι πολύ σημαντικός εταίρος για όλους μας. Ειδικά αυτούς, αυτή την χρονική στιγμή που ζούμε σε ένα πλαίσιο κρίσης με την Ουκρανία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πέτερλε για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ πραγματικά θα λυπηθώ Α, αν είναι αυτή η τελευταία έκθεση της ε, κυρίας Σόμαν Ρόιτεν για την Τουρκία. Μας είχε καλομάθει στην ποιότητα και ήταν πραγματικά ισορροπημένες οι εκθέσεις ε, και θέλω να την ευχαριστήσω ακόμη μια φορά, να γνωρίζει την πρόοδο που υπάρχει, ασκεί κριτική όπου πρέπει. Εγώ δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, θα κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Η διαδικασία αυτή διαπραγματεύσεων λαμβάνει χώρα σε ένα πάρα πολύ περίπλοκο πλαίσιο οι πολιτικές διαφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη η ε, τα πολιτικά γεγονότα στην Τουρκία και στον ευρύτερο χώρο και διαπιστώνουμε πως ε, η διαδικασία αυτή οδήγησε σε κάποιες μεταρρυθμίσεις ε, και βεβαίως είναι απαραίτητη για την περαιτέρω πρόοδο της Τουρκίας και θα ήθελα να αναφερθώ στο λεγόμενο δημοκρατικό πακέτο παρά το ότι βεβαίως δεν ε, υπάρχει αρκετή προσοχή για τους αλεβίτες. Ε, παρά το ότι η έκθεση βεβαίως αφορά το 2013 θα ήθελα να πω πως προσεχω... Ε, προσφάτως με συγχωρείτε πέρασε το πέμπτο πακέτο της δικαιοσύνης που αφορούσε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επίσης σε λίγο καιρό θα έχουμε και την απελευθέρωση της ε, βίζας. Αλλά βεβαίως υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα με την διαφθορά, το πώς καθορίζεται η συνωμοσία και βεβαίως η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο σε όσους έχουν ζητήσει στη διαδικασία του ΚΑΤΣΔΙ. Ο κύριος ε, Κόρκολα. Κυρία Κορκόλα, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Σήμερα μάθαμε ότι υπήρξε ένα νέο θύμα. Αυτός ο 15χρονος ε, έφηβος ε, κατέληξε. Στην ε, έκθεση προόδου για την Τουρκία Μιλάμε φυσικά για παραβιάσεις της ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συνολικά αυτό που έγινε στον Κεζί είναι ένα μέρος μόνο, αλλά δεν θέλω να τα ξεχνάμε όλα αυτά. Επίσης με ανησυχεί η δήλωση του κυρίου Ερντογάν, σύμφωνα με την οποία δεν θα σεβόταν την υπόσχεσή του να μην διεκδικήσει ε, για τέταρτη φορά την εξουσία, από ό,τι φαίνεται δεν θα σεβαστεί πια τις υποσχέσεις του και έχουν γραφτεί πάρα πολλά για αυτή την ασθένεια των δεκαετών, δηλαδή η εξουσία ρωσταίνει τους ανθρώπους. Εγώ νομίζω ότι ο Ερντογάν θα πρέπει να αποχωρήσει πλέον και αυτό θα είναι καλό για την προσχώρηση της Τουρκίας. Σας ευχαριστώ, ο κύριος Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω πως η συζήτηση σήμερα το βράδυ είναι κάπως σουρεαλιστική γιατί νομίζω ότι εδώ κάνουμε τον χώρο των υποκριτών. Τι ακούμε εδώ και μία ώρα. Κάποιες αρνητικές αξιολογήσεις για την τρέχουσα κατάσταση στην ε, Τουρκία. Τη δικαστική, την πολιτική, την επιχειρηματική, της παιδείας, ε, του σεβασμού των ε, θρησκευτικών μειονότητων, όλα αρνητικά. Και τι προτείνουμε στην έκθεση. Να ανοίξουμε για άλλα κεφάλαια. Άρα λοιπόν αυτή η εντύπωση ότι ανοίγοντα κεφάλαια διαπραγματεύση θα επηρεάσουμε ουσιαστικά την κατάσταση είναι ο λάθος δρόμος. Χρειαζόμαστε μια πολύ πιο απαιτητική προσπάθεια πολιτικού διαλόγου με την Τουρκία, με την Τουρκία που είναι μεγάλος εταίρος, αλλά το να ανοίξουμε διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή ανταμείβει ένα τουρκικό καθεστώς το οποίο κάνει λάθος βήματα. Άρα λοιπόν για το κεφάλαιο 23 να μου πει θα το ανοίξουμε, το θέλουν οι Τούρκοι. Μα με συγχωρείτε, εμεί εδώ δεν μα έστειλαν ούτε οι Τούρκοι ούτε εκπροσωπούμε του Τούρκου. Οι Ευρωπαίοι πολίτε μα έστειλαν εδώ και δεν είμαι σίγουρη ότι θέλουν να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Συνάδελφο Λούτσεβα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συζητάμε μια έκθεση που έχει να κάνει με τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και ανησυχώ ιδιαίτερα από το γεγονός ότι αν στις Βρυξέλλες ε, εκφράζουν τις επιθυμίες τους ε, για την καλή γειτνίαση οι Τούρκοι ε, ταυτόχρονα στέλνουν και ε, αντιφατικά μηνύματα. Η έκθεση λέει ότι έχει συμμορφωθεί η Τουρκία με τις διεθνείς συμβάσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί η Τουρκία συνεχίζει να μη σέβεται τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει έναντι της Βουλγαρίας βάσει της συμφωνίας της Άγκυρας για τη χορήγηση αποζημιώσεων ε, στους Βουλγαρούς από την περιοχή της Θράκης και επίσης επίσης δεν έχει υπάρξει πρόοδος από το 2008. Πρόκειται για ένα κενό στην τουρκική πολιτική που πρέπει να καλυφθεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να υπερασπίσει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συνάδελφο Σπίτσουλα. Η Τουρκία είναι ένας πιθανός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για το λόγο αυτό οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να συνεχιστούν άσχετα με το πόσο χρόνο θα χρειαστούν. Η κατάσταση με τις διαπραγματεύσεις περιγράφεται σωστά και όλα τα κράτη τα οποία βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να εκπληρώσουν τα ίδια κριτήρια. Και νομίζω ότι τα αποτελέσματα από την από 9 χρόνια, ε, τα αποτελέσματα είναι μάλλον πτωχά. Κακό αυτό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Τουρκία. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να δούμε ποια είναι τα κομμάτια που μας ενδιαφέρουν όλους και τις δύο πλευρές, δηλαδή ασφάλεια, εμπόριο κτλ. Και να εστιάσουμε εκεί, γιατί αυτή τη στιγμή πάνω από μισό εκατομμύριο ε, πρόσφυγες από τη Σερβία είναι στην Τουρκία. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει εμείς να δούμε τα θέματα αυτά. Μην ξεχνάτε πως υπάρχει το θέμα της Κύπρου ε, και δεν θα πρέπει να απομονώσουμε τους ε, Τουρκοκυπρίους. Επίσης υπάρχει και το θέμα των θεωρήσεων με την Τουρκία και αυτό μην το αφήνετε στην άκρη. Ε, Ευχαριστώ κύριε Παπαδοπούλου. Κυρία Πρόεδρε, όσον και αν επιχειρείται από ενοχοποίηση της Τουρκίας και ωρεοποίηση του ρόλου της, τα γεγονότα βοούν σκάνδαλα, διαφθορά, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων μη τήρηση των κριτηρίων της κοπεγχάγης η έκθεση δυστυχώς περιορίζεται σε παρενέσεις δεν επιβάλλει κυρώσεις. αντίθετα επιδιώκει να επιβραβεύσει την τουρκική θρασίτητα αφού καλεί για άνοιγμα των κεφαλαίων 23-24 χωρίς η τουρκία να έχει εφαρμόσει το πρωτόκολλο της άγκυρας χωρίς να έχει υπογράψει τη σύμβαση του ΟΕΕ εθνών για το δίκαιο της θάλασσας χωρίς να έχει τερματίσει την κατοχή της κύπρου. ζητά άνοιγμα του κεφαλαίου 15 για την ενέργεια αγνοώντας τις τουρκικές τουρκικέ απειλέ και την παρουσία των τουρκικών σκαφών ύβρο και μπαρπαρός στην κυπριακή ναός η τουρκία κρατά την αμόχωστον υπομοιρία ζητώντα ανταλλάγματα και απευθεία εμπόριων αντί να εφαρμόσει το ψήφισμα 550 του οργανισμού ηνωμένων εθνών. συνεχίζει τον παράνομο επικισμό και την καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων προσφύγων αγνωμένων και εγκλωβισμένων στην κύπρο. κύριε φούλε η τουρκία παραβιάζει το διεθνέ δίκαιο και όμω παραμένει ατιμόρυτη. αυτό εξευτελίζει την ίδια την ευρωπαϊκή ένωση το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις αρχές για τις οποίες όλοι έπρεπε να σεβόμαστε και να παλεύουμε. δυστυχώς η ευρωπαϊκή ένωση επιβραβεύει την τουρκία αντί να την τιμωρεί. επιτέλους ας το αντιληφθούμε. Ευχαριστώ. Η συνάδελφο Σιράτση Πολυπετία. Ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω ε, να υπογραμμίσω μία πτυχή που πρέπει να επισημαίνουμε στο κείμενο. Το θέμα της επίλυσης του Κουρδικού δεν είναι δυνατή η προσχώρηση της Τουρκίας χωρίς να έχει επιληθεί το κουρδικό ζήτημα δημοκρατικά ε, ε, στέλνουμε τεράστιο μήνυμα στον πληθυσμό, γι' αυτό πρέπει να προωθήσουμε την ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ του ΠΚΚ και των τουρκικών αρχών. Πρέπει να γίνουν σεβαστές οι δεσμεύσει. Το ΠΚΚ πρέπει να εγκαταλείψει τα όπλα και να ε, προχωρήσει προς την ειρηνευτική διαδικασία και θα πρέπει η κουρδική κυβέρνηση να διασφαλίσει την εκπαίδευση στην κουρδική γλώσσα, η αναγνώριση της κουρδικής ταυτότητας ε, και τη ε, μειονότητας στο σύνταγμα Σύνταγμα και τέλος να ε, καταργήσει τον εκλογικό νόμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Τόμασιτς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η συζήτηση για την θέση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχιστεί βεβαίως, αλλά πέραν από το ευρωπαϊκό μέλλον τη ε, γεγονός είναι πω πρέπει να συνεργαστούν ε, Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία βρίσκεται στα εξωτερικά μας σύνορα, είναι σύμμαχος μας στο ΝΑΤΟ και πολλοί Ευρωπαίοι κατάγονται από την Τουρκία. Αλλά εγώ θα ήθελα να τονίσω μια άλλη πτυχή, τους δεσμούς ε, οι οποίοι επιβάλλουν ευθύνες και στις δύο πλευρές και θα ήθελα να τονίσω μία πτυχή μόνο. Το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, ειδικά το εμπόριο λαθρεμπόριο ηρωίνης από το Αφγανιστάν. Η Κροατία βρίσκεται στον λεγόμενο δρόμο των βαλκανικών των ναρκωτικών και παρά το ότι η Τουρκία πιάνει μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών κάθε χρόνο δεν επαρκεί αυτό. Πρέπει να δώσει βάρος στον τομέα αυτό, πρέπει να αδανοποιηθεί αυτός ο δρόμος και να ενταθεί ο αγώνας κατά των ναρκωτικών. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνει τη διαδικασία Κατστιάη. Και τώρα το λόγο έχει επίτροπος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμο μέλη. Προεδρία. Για την Τουρκία πάντοτε ετοιμάζω κάποιες καλές δηλώσεις, αλλά σπανίως τις χρησιμοποιώ. Γιατί η συζήτηση πάντοτε με κάνει να σκέφτομαι πώς να αντιδράσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτό το ευρύ φάσμα των απόψεων. Καθώς είναι λοιπόν τα τελευταία μου σχόλια ε, σε αυτή τη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο και έχοντας αυτή τη θέση θα σας παρουσιάσω μια πιο προσωπική άποψη. Θα αναφερθώ σε τρία σημεία. Το πρώτο. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να γίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Τουρκία να σεβαστεί όλες τις υποχρεώσεις που έχει για όλα τα κεφάλαια της προσχώρησης. Δεν υπάρχει παρέκκληση από το σεβασμό των θεμελιωδών ευθεριών, του κράτους δικαίου, τη λογοδοσία και την διάκριση των εξουσιών. Δεν υπάρχουν ε, ενδιάμεσες ε, περίοδοι, δεν ε, υπάρχουν παρακάμψεις που θα αγνοούσαν αυτή τη διαδικασία της προσχώρησης ε, όπου η πολλαπλή συμμόρφωση είναι το κύριο μας εργαλείο. Και αυτό που πάντοτε ανέμενα από αυτό τον Νίκο είναι να θέσει το σωστό ερώτημα και να μου βοηθήσει να βρω τη σωστή απάντηση. Όμως, δεν θα βοηθήσετε εμένα, θα βοηθήσετε το διαδοχό μου. Αν συνεχίσετε να λέτε ότι θα πρέπει να είμαστε πιο πατητικοί, Αφενός. Αλλά και πιο περιοριστικοί ως προς ε, την έναρξη των ε, διαπραγματεύσεων προσχώρησης. Γιατί σε αυτό θα μπορούσα πράγματι να απαντήσω την πιο σχετική ερώτηση και την άκουσα μία-δύο φορές στο παρελθόν, όχι στην πραγματικότητα σήμερα. Και είναι, θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να αποτελεί κριτήριο αναφοράς για τις μεταρρυθμίσεις της Τουρκίας ή όχι. Αυτή είναι η ερώτηση. Δεύτερον, δεν υπάρχει άλλος τρόπος κανένας άλλος τρόπος ε, να λύσουμε συνολικά το κυπριακό ζήτημα παρά με βάση τις ευρωπαϊκές αξίες. Και χαίρομαι που βλέπω ότι και με την τουρκική εμπλοκή μπορέσαμε να δούμε, να σημειώνεται πρόοδος ε, σε αυτό το θέμα. Μόλις σήμερα Δύο συνομιλητές ε, συναντήθηκα στην προστατευμένη περιοχή των Ηνωμένων Εθνών και θα συνεχίσουν τις συζητήσεις ε, την Παρασκευή 14 Μαρτίου. Σήμερα επιβεβαίωσαν ε, ότι στις 31 Μαρτίου 2014 θα συναντηθούν και οι ηγέτες. Και υπάρχει και ένα τρίτο στοιχείο. Ένα νερό, ένα νερό αγόρι 15 ετών. Αναφερθήκατε πολύ σε αυτόν μετά από 260 μέρες ε, σε κόμμα. Τυπήθηκε από ένα δακρυγόνο που έριξε η αστυνομία κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης. Είναι πάρα πολύ λυπηρό αυτό το γεγονό. όμως μας υπενθυμίζει τις φιλοδοξίες ε, του λαού της Τουρκίας εγώ έχω ακούσει αυτές τις προσδοκίες και πάντοτε θα με καθοδηγούν στις προσπαθίες μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κουρκούλας έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ το Σώμα για την ενδιαφέρουσα συζήτηση η οποία πιστεύω δείχνει ξεκάθαρα πόσο αναγκαίο είναι να συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε τις πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις στην τουρκία. Αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε μπροστά και πρέπει να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. όπως άλλωστε επισημαίνει και το ψήφισμά σας όλες οι πλευρές έχουν πολλά να κερδίσουν από την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις και από την περαιτέρω πολιτική μεταρρυθμίσεων πολιτικών και οικονομικών στην τουρκία από πλευρά μα η προεδρία μαζί με τα κράτη μέλη και την επιτροπή κάνουμε ό,τι δυνατόν για να σημειωθεί πρόοδο. η τουρκία είναι σημαντικό εταίρο τη ευρωπαϊκή ένωση και η πρόοδο στην προσέγγιση τη με την ευρωπαϊκή ένωση είναι και θα είναι προ όφελο όλων. βεβαίω το άνοιγμα διαπραγματευτικών κεφαλαίων δεν είναι αυτό ο σκοπό. είναι η κατάληξη το επιστέγασμα μια διαδικασία η τουρκία γνωρίζει καλά τι πρέπει να πράξει και στον τομέα αυτό. το έχει συζητήσει επανειλημμένως με την επιτροπή με το συμβούλιο στο πλαίσιο του συμβουλίου σύνδεσης αλλά και σε διμερές επίπεδο με τα κράτη μέλη. το ζητούμενο συνεπώς είναι η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για την οικοδόμηση κράτους δικαίου και το σεβασμό στην πράξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων καθώς επίσης και η υλοποίηση των διεθνών υποχρεώσεων της τουρκίας. η διεύρυνση είναι διακυβερνητική διαδικασία. η πρόοδος εξαρτάται κυρίως από την τουρκία και δεν πρέπει να παροράτε ότι στην περίπτωση της τουρκίας το άνοιγμα και το προσωρινό κλείσιμο κεφαλαίων υπόκειται επίσης και στα συμπεράσματα του συμβουλίου της 11 η Δεκεμβρίου του 2006. Θα ήθελα ανακεφαλαιώνοντας να υπενθυμίσω ότι εν τέλει αυτό που θα καθορίσει το ρυθμό των διαπραγματεύσεων είναι η ικανότητα της ίδιας της τουρκίας και η βούλησή της να προχωρήσει. η προώθηση των διαπραγματεύσεων θα απαιτήσει όχι μόνο γενικές περαιτέρω μεταρρυθμίσεις και προσπάθειες μεταρρυθμίσεων αλλά και θαραλέες πολιτικές αποφάσεις από πλευράς τουρκίας. από πλευράς μας θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. τέλος θα ήθελα να επισημάνω τη σημασία του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και της εμπλοκής του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου για την ευρύτερη πολιτική διαδικασία εντός της οποίας λειτουργούμε. η δέσμευση των πολιτών της τουρκίας και των κρατών μελών της ευρωπαϊκής ένωσης στη διεξαγωγή δημοκρατικού διαλόγου έχουν κέρια σημασία για τη διασφάλιση συνεχούς υποστήριξης σε αυτή τη σπουδαία ιστορική διαδικασία μεταξύ τουρκίας και ευρωπαϊκής ένωσης. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι έχω λάβει μια πρόταση ψηφίσματος. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο, Τετάρτη, 12 Μαρτίου, στις 12 το μεσημέρι.